τι μεγαλύτερε πολιτιστικέ αξίε που έχει ο κάθε πολιτισμό και να αφήσουμε τα αρνητικά πίσω μα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε την ε, ε, τόλμη να πούμε ότι δεν μπορεί η βία να δικαιολογείται από την παράδοση, την ιστορία, τη θρησκεία. Ε, όχι, ψάχνουμε οικουμενικέ αξίε που έχουν ήδη καταγραφεί ούτω ή άλλω στην Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών και θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφεί προ αυτό. Επίση, θα πρέπει η πολιτιστική, μάλλον η κουλτούρα ως προς τα θέματα αυτά, η νοοτροπία να αλλάξει και να υπάρξουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης ε, για τα δικαιώματα των γυναικών. Όπως προσπαθεί να κάνει το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και πολλές ενώσεις των γυναικών στα κράτη-μέλη μας. Πρέπει να συνεργαστούμε με επαγγελματίες σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η πρόληψη, οι κοινωνικές υπηρεσίες προκειμένου να εντοπίσουμε καλύτερα τις ομάδες που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο και να μπορέσουμε να προσφέρουμε πρόληψη, μέτρα πρόληψης Πρόεδρε, εγώ συμμετείχα στην εκστρατεία που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μηδενική ανοχή κατά του ακροτηριασμού των γυναικείων γενετικών οργάνων και ελπίζω ότι όλοι θα δεσμευτούμε στον αγώνα αυτό και θα ε, επιδιώξουμε μαζί έντονη δράση. Ε, πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Γκουρμάη. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Παρόλο το, παρά το γεγονό ότι το φαινόμενο αυτό αναγνωρίζεται περισσότερο από τη Διεθνή Κοινότητα Υγεία και του ε, εντυπωσιακού αριθμού, το φαινόμενο παραμένει σχετικό εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται μόνο για σοβαρή παραβίαση των, κατάφορη παραβίαση των βασικών δικαιωμάτων ε, γυναικών και κοριτσιών, αλλά πραγματικά θέτει σε κίνδυνο την υγεία των γυναικών και τι ε, εμποδίζει να ασκήσουν τα βασικότερα δικαιώματά του. Η βάρβαρη αυτή πρακτική λοιπόν, λοιπόν, επειδή ακριβώ συμβαίνει πολλέ φορέ εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ δύσκολο να αντιπιστεί και θα πρέπει να αναλάβουμε δράσει εκπαίδευση και ενημέρωση ε, για όλου του ενδιαφερομένου. Τα προγράμματα που έχει επιχειρήσει ω τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τη UNICEF έχει επιτρέψει να υπάρξουν κάποια πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Αλλά τώρα που να εντείνουμε τι προσπάθειέ μα για την εξάλληψη του κατηρισμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, πρέπει να προβλέψουμε ένα ευρύτερο ε, πρόγραμμα δράση για την αντιμετώπιση τη βία λόγω του φύλου θα πρέπει να υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζω το γεγονό ότι το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων ε, προβλέπει την ε, συγκέντρωση δεδομένων για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σκληροί ε, ω προ του προμηθευτέ υπηρεσιών υγεία που θα επιτρέψουν τέτοιου είδους πρακτικές βάσει της αρχής της ε, εξωταθικότητας που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάποια κάτι μέλη. Και θα πρέπει ακόμη και ε, στα σύνορά μας να λάβουμε μέρημνα για τις κοινότητες που ενδεχομένως να κατοικούν εκεί. Πάντως, μια και είναι εδώ επίτροπος, να τον ευχαριστήσω για το εξαιρετικό του έργο. Ελπίζουμε να είναι πάλι στη θέση του και μετά, γιατί χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους σε τέτοιες θέσεις. Ευχαριστούμε κυρία Λάτφορντ. Um, Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μεγάλη μου χαρά συμμετέχω σε αυτή τη ε, διακομματική συζήτηση και ε, χαίρομαι που εγκαταλείψαμε αυτό. Μάλλον όλοι συμφωνούμε ότι όταν μιλάμε για κλειτοδεκτομή πρόκειται για μια βάρβαρη πρακτική. Ε, ο γυναικείος ο ακροτηριασμός των γυναικείων γενικών οργάνων δεν λέει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ένα βασανιστήριο. Ε, κατά των γυναικών και των παιδιών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε 25-65.000 γυναίκε που πλήττονται από αυτού του είδου την πρακτική. Είναι 65.000 οι γυναίκε που μπορεί να βρισκόνται σε κίνδυνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει ε, να, μην, να υπάρξει μηδενική ανοχή για τέτοιου είδου ε, φαινόμενα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η δίωξη μπορεί να εφαρμοστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει των στοιχείων που έχουμε, αλλά ισχύει ω αδίκημα αυτό θεωρείται έγκλημα εδώ και ε, δεκαετίες. Δεν υπήρξε καμία επιτυχη δίωξη. Και οι ιδιοκτικέ μας αρχές που αυτή τη στιγμή στις οποίες ηγείται μια γυναίκα έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο γυναικών ε, σε όλη τη χώρα που παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου αλλά πρέπει περισσότερο να δώσουμε έμφαση στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση. Ε, πραγματικά χρειάζεται εδώ μια ευρωπαϊκού επίπεδου πρωτοβουλία. Χαίρομαι που η υπουργό που είναι υπεύθυνοι για την ανθρώπινη ανάπτυξη στον Ηνωμένο Βασίλειο ε, από το κόμμα μου έχει ε, προβλέψει 35 εκατομμύρια ε, βρετανικές τερλίνες ως κονδύλι διεθνώς για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο αυτό και σήμερα το μεσημέρι 11 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου θα υπάρξει μια εκδήλωση για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού διεθνώς. Σας παρακαλώ να συμμετάσχετε. Κυρία Μπόερ, για να μην Μπάουερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Τι δείχνει η σημερινή συζήτηση. Ε, τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Ακούσαμε ότι πρόκειται για 140 εκατομμύρια γυναικών και πλέον που έχουν υποστεί αυτή τη βία. Η Αίγυπτος, Αιθιοπία, Σομαλία και Σουδάν είναι οι χώρες όπου απαντά περισσότερο. Ο επιπολασμός εκεί μπορεί να είναι μέχρι και 98%. Σε άλλες χώρες όπως η Νιγηρία, Κένια, τον Κόσενα, Γάλλη, ο επιπολασμός ε, κυμαίνεται 30 με 50%. Δεν υπάρχει όμως μόνο στην Αφρική αυτό το φαινόμενο και σε τμήματα της Μέσης Ανατολής, Ομάν, ε, η Εμένη στο Ιρακινό Κουρδιστάν και μεταξύ ορισμένων γυναικών Βεδουίνων ακόμα και στο ίδιο το Ισραήλ. Οι στατιστικές που πρόσφατα εξέδωσε η UNICEF και αναλύουν ε, στοιχεία από 29 χώρες στην Αφρική ε, δείχνουν ότι 18 από 29 χώρες είναι στη Δυτική και Κεντρική Αφρική και το φαινόμενο αφορά το 1 πέμπτο των ε, κοριτσιών στην υποσαχάρια Αφρική. Αυτός ο ακροτηριασμός γίνεται κυρίως ε, κορίτσια πολύ νεαρά, από βρέφη μέχρι 15 ετών και πρόκειται για σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών και βία κατά των κοριτσιών και γυναικών πολύ ε, βαριά ταυτόχρονα. Ε, επειδή έχουμε και πρόσφυγες και μετανάστες και αντίστοιχα ρεύματα, Εμφανίζεται και αλλού αυτό το φαινόμενο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως ακούσαμε υπολογίζεται σε 500.000 ο αριθμός των γυναικών στην Ευρώπη. Δέκα είναι τα κράτη-μέλη που έχουν ειδικέ διατάξεις στο ποινικό τους δίκαιο για τον ακροτηριασμό, αλλά βάσει ε, των ποινικών ε, κωδίκων μπορεί να διωχθεί ως κακούργημα σε όλα τα κράτη-μέλη. Αναγνωρίζεται σε αυτό και η ετεροδικία. Σε 13 κράτη-μέλη, ακούσαμε, στη Γαλλία υπάρχουν ε, πάνω από 60.000, στο Ηνωμένο Βασίλειο πάνω από 65.000 γυναίκες. Και όπως ακούστηκε επίσης, παρά το γεγονός αυτό, η καταστολή και η δίωξη δεν βοηθάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σπάνια. Ε, αυτό που χρειαζόμαστε είναι πραγματικά επιβολή του νόμου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκαρσία Πέρες, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο ακροτηρισμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και σαφή και κατάφορη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων ήταν απαραίτητο να αποφανθεί το Κοινοβούλιο κατά αυτού του φαινομένου. Μιλήσαμε για δεδομένα, στοιχεία. 140 εκατομμύρια γυναικών και κοριτσιών σε όλο τον κόσμο, 500.000 στην Ευρώπη. Υπάρχουν μελέτες που λέγουν ότι ε, περίπου 17.000 κορίτσια στη χώρα μου, την Ισπανία, κινδυνεύουν να πέσουν θύματα αυτού του ακροτηριασμού. Θα πρέπει λοιπόν με ικανοποίηση να υποδεχθούμε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να καταλάβουμε ότι είναι απαραίτητο πλέον να περάσουμε από τα απλά λόγια στα ουσιαστικά έργα. Σε δράση να προωθήσουμε διάφορες στρατηγικές ε, υπέρ της πρόληψης και της εξάλληψης αυτού του ακροτηριασμού που είναι ομή και κατάφορη βία κατά των γυναικών. Είναι απαραίτητο να επιμείνουμε στη σημασία ε, της εκπαίδευσης των υγειονομικών, των γιατρών και γενικότερα ε, της παιδείας. Συνεργασία μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών που εργάζεται στην κατεύθυνση αυτή για να τερματιστεί αυτή η βία που δεν χωράει στον 21ο αιώνα γιατί αν κάποιος ισχυρίζεται ότι δικαιολογείται αυτό ε, βάσει κάποιων δικαιολογιών να πούμε ξεκάθαρα ότι ο σεβασμός στην παράδοση και στον πολιτισμό έχει μια κόκκινη γραμμή απαραβίαστη που είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το λόγο έχει η κυρία Χόλ για να μην Πρόεδρε, και εγώ καλωσορίζω τους Βρετανούς συνοδέλφους, μάλλον την ε, πρωτοβουλία της Βρετανής Υπουργού, ε, της κυρίας ε, Φέδεστον, να φέρει την προσοχή, να προσελκύσει την προσοχή για το φαινόμενο αυτό και να το θέσει ως προτεραιότητα και για μας, για τη χώρα μας και για τις υπόλοιπες. Θα πρέπει λοιπόν η ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κάτι μέλη να συνεργαστούν και να προβλέψουν κονδύλια για την αντιμετώπιση αυτής της πρακτικής. Διότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να αναλάβουμε μέτρα στις τοπικές κοινότητες. Όταν οι οικογένειες δημοσίω μπορούν να παραδεχτούν ότι έχουν εγκαταλείψει την πρακτική του ακροτηριασμού τότε μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Όμως, ε, πέραν της πραγματικής ε, αντιμετώπισης σε τοπικό επίπεδο, θα πρέπει και σε διπλωματικό επίπεδο να υπάρξει πρωτοβουλία, ώστε με τους Αφρικανούς εταίρους μας να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για να υπάρξει μια κοινή συνεννόηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Τον επόμενο μήνα, εδώ στο Στρασβούργο, η κοινή κοινοβουλευτική συνέλευση θα συνέλθει και θα ήθελα εδώ να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι ειδικές έχει ε, προβλέψει, έχει προγραμματίσει για να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία τη συνάντηση αυτή ώστε να πιέσει να υπάρξει κοινή δράση ε, μεταξύ ε, Ευρώπη και Αφρικανικών ε, χωρών ώστε στην πράξη να υλοποιηθεί η δέσμευση να αναχαιτιστεί το φαινόμενο αυτό του ακροτηρισμού των γυναικείων γενικών οργάνων και να εξαλειφθεί μια για πάντα. Πρόκειται για παραβίαση δικαιωμάτων του παιδιού και πρέπει να πάυσει. Ευχαριστούμε η κυρία Ματέρα για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε συνάδελφοι, σήμερα θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Διότι όταν μιλάμε για ακροτηριασμό των γυναικείων γενετικών οργάνων, μιλάμε για βία κατά των γυναικών. Το κοινοβούλιο αυτό ήδη το 2009 εκφράστηκε με την πλειοψηφία του εγκρίνοντας έκθεση πρωτοβουλίε ακριβώς για το θέμα αυτό, αλλά και πάλι σήμερα το θέμα αυτό δεν αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για περίπτωση αδράνειας, πρόκειται για έναν κόλαφο κατά των δικαιωμάτων των γυναικών με, 50, με 55 εκατομμύρια γυναίκες ε, ε, στο, στην Επιρώ που έχουν υποβληθεί στην πρακτική 125 διεθνώς και ε, ένα κορίτσι κάθε 6 λεπτά που ακροτεριάζεται διεθνώς και πραγματικά αποδεικνύει ότι η Ευρώπη δεν είναι το λίκνο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαι υπερήφανη που η χώρα μου έχει προβλέψει ειδική νομοθεσία εξαιρετικά εξελιγμένη με νόμο του 2006 όπου απαγορεύεται ο ακροτηριασμός των γυναικείων γενετικών οργάνων σε όλη τη χώρα προβλέποντας την πρόληψη πολυάριθμων δράσεων αντιμετώπισης και ενημέρωσης για αυτού του είδους την απαράδεκτη μορφή βίας. Ιδού συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, νομίζω το πιο σημαντικό που έχουμε να πούμε, το πιο ισχυρό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας είναι η πρόληψη, αντιμετώπιση, αναχέτηση και πρόληψη. Και για άλλη μια φορά είμαι πολύ ικανοποιημένη γι' αυτό. Με 4 εκατομμύρια ευρώ η χώρα μου, ένα κονδύλι σίγουρα όχι θεαματικό, αλλά τουλάχιστον σημαντικό, έχει προβλέψει να εκτελέσει μια ενημερωτική εκστρατεία που ονομάζεται «Εκανής ε, εκτός» μια εκστρατεία που θα ενημερώσει γονείς ε, και δασκάλους για την ε, ανάγκη να πάυσει η πρακτική αυτή ε, του ακροτηριασμού στα κορίτσια και υπάρχει και ένα δωρεάν νούμερο που μπορεί να δώσει, κανείς, να δώσει πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερο για το φαινόμενο αυτό στην Ιταλία. Θα πρέπει λοιπόν στην Ευρώπη να επικεντρωθούμε στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, να κοιτάξουμε πώς θα υλοποιήσουμε και θα στηρίξουμε το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ακριβώς για το θέμα αυτού του κριτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Η αδράνεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώ έλλειψη ανάληψη δράση. Ένα θέμα που τόσο πολύ αφορά όλε μα, αλλά είμαι βέβαια αφορά και του άντρε. Τη βία δηλαδή κατά των γυναικών. Ευχαριστούμε την κυρία Ματέρα και κυρία Κοστέλο. Επειδή σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα για την καταπολέμηση του γάμα α, πρέπει και εμείς να το γιορτάσουμε στο Κοινοβούλιο. Το γάμα σίγμα α είναι τρομακτική πρακτική. Εκατομμύρια γυναικών, δύο εκατομμύρια το χρόνο υποβάλλονται σε αυτή την πρακτική. Και στη χώρα μου πάνω από 3.500 γυναίκες έχουν υποβληθεί σε γάμα σίγμα α. Και πολλές φορές πρόκειται για κορίτσια, επομένως πρόκειται για βιοπραγία κατά των παιδών. Το πρόγραμμα δράσης της Κομισιόν είναι μια καλή αρχή και βάση για περαιτέρω δράση ανάλογη με εκείνη που είχε αναλάβει προηγουμένως η Διεθνής Αμνηστία. Οι προσπάθειες που είχαν γίνει για την κατάργηση του ΓΣΑ σημείωσαν τελευταία, μια τελευταία επιτυχία και στη Σομαλία. Πρέπει όμως να μιλήσουμε και για την πρόληψη, για την αλλαγή νοοτροπίας. <clears throat> Γιατί το γάμα σίγμα αλφα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο θρησκευτικά. Υπήρξαν και άλλα ψηφίσματα της Αφρικανικής Ένωσης ας πούμε καταδίκης του γάμα σίγμα αλφα και χαίρομαι ιδιαίτερα Επίτροπε που λέτε ότι και η Ένωση θα συνεχίσει να το πιέζει το θέμα με την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Στη Σομαλία θα αναλυφθεί τον επόμενο μήνα η επόμενη εκστρατεία. Πρέπει η κοινωνική λειτουργή και οι δάσκαλοι να έχουν συνείδηση του γεγονότος και του φαινομένου για να υποστηρίξουν τις σχετικές αιτήσει και την καμπάνια και παρακαλώ και τους βουλευτές να την υποστηρίξουν. Ευχαριστούμε κυρία Κοστέλο και κυρία Μωρέν Σαρτιέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εδώ αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να συζητήσουμε γιατί είναι αντίθετο με όλες τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα δε την ισότητα των πολιτών, την ισότητα των φίλων και την προσάσπιση των γυναικείων δικαιωμάτων καθώς και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Δεν άκουσα όμως ούτε έναν σήμερα να διαφωνεί. Έχουμε το κείμενο, τη χάρτα των θεμελιωδών, τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ξέρουμε όμως πόσα θύματα κλειτοριδεκτομών σημειώνονται, πόσοι ακροτηριασμοί πόσους ακροτηριασμού υφίστανται οι γυναίκες δεν το ξέρουμε ακριβώς. Οι σεξουαλικοί ακροτηριασμοί είναι μία τρομακτική μείωση της αξιοπρέπειας των γυναικών και κοριτσιών και νέων κοριτσιών διότι ο, η κλειτοριδεκτομή γίνεται σε πολύ νεαρή ηλικία. Πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθούμε για τα ανυπεράσπιστα αυτά κοριτσάκια. Πρόκειται για πολιτιστική πρακτική αλλά και πέρα από αυτήν για βάρβαρη πρακτική. Οι ακροτηριασμοί αυτή είναι οριστική. για όλη τη ζωή της γυναίκας. Είναι πρόβλημα υγειονομικό, υγείας, υγιεινής και μπορεί και να οδηγήσει στο θάνατο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοια πράγματα. Γίνονται και μέσα στην Ένωση και εκτός και δεν δικαιολογεί αυτό ότι δεν είμαστε ε, υπεύθυνοι. Πρόκειται για τρομερή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάζει το δικαίωμα στην υγεία, στην ασφάλεια, στη σωματική ακαιρεότητα και στην μη υποβολή σε βασανιστήρια. Η Γαλλία ήταν από τις πρώτες χώρες που χορηγούσε άσυλο σε γυναίκες που έχουν υποστεί γάμα σίγμα αλφα. Και σκοπεύουμε να εγκρίνουμε και ένα σχετικό νόμο. Τα πολιτιστικά αυτά προβλήματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και με τους, σε συνδυασμό και με τους άντρες και με τα αγόρια με καμπάνιες πληροφόρησης φυσικά και προς τις νεαρές γυναίκες και τα κορίτσια καμία παράδοση δεν μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη και θεμητή με τέτοιου είδους βάρβαρες πρακτικές και γι' αυτό θα ήθελα και στην παράγραφο 4 που ζητάμε πραγματικά πανενωσιακή νομοθεσία να εφαρμοστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μωρέν Σαρτιέ. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαιρόμαστε εδώ και συγχαίρουμε ένα τον άλλον για τη σημερινή ημέρα. Εγώ δεν έχω να συγχαρώ κανέναν. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε χρόνο που περνάει θα πρέπει να είναι διεθνή ημέρα κατά του ακροτηρισμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Έχω συμπληρώσει 15 χρόνια εδώ μέσα και δεν μπορώ να πιστέψω ότι ακόμα καθόμαστε εδώ και στεκόμαστε και ζητούμε δράση. Ωραία η ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει ε, έξι γενικέ διευθύνσει να ασχολούνται γιατί είναι εργάστιο το, θέμα, εγκάρσιο οριζόντιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρειαζόμαστε πρόγραμμα δράσης πριν λήξει η θητεία σας. Ε, ο ακροτηριασμός αυτός ε, έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως παραβίαση των ανθρωπίνων, γυναικείων, παιδικών δικαιωμάτων και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο εάν καταλάβουμε ότι έχουν συνολικά δικαιώματα οι γυναίκες. Αυτό ε, συμπεριλαμβάνει και τα δικαιώματα τα σεξουαλικά, της υγείας, της αναπαραγωγικής υγείας. Και δεν θα πρέπει να αποφασίζει ένας άντρας και ακόμα λιγότερο ένας κληρικός τι θα κάνει μια γυναίκα το σώμα της. Έχω δει εγώ τις σωματικές επιπτώσεις αυτού του ακροτηριασμού και είναι τρομακτικές, φρικτές. Τώρα έχει έρθει η ώρα για δράση. Τα στοιχεία, οι αριθμοί ε, μας τρομοκρατούν στα κράτη-μέλη. Ε, και κύριε Επίτροπε, ακούστε με γιατί ξέρω ότι ακούτε. Θα πρέπει να απευθυνθούμε στους φίλους μας και εκείνους που δεν θέλουν να το αντιμετωπίσουν πρόσωπο με πρόσωπο περισσότερη δράση, λιγότερα λόγια. Γι' αυτό καλό όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης να προσυπογράψουν την ε, Σύμβαση για την ε, καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Χρειαζόμαστε αυτό το ευρύ πλαίσιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω να μην ξανασυζητήσουμε ποτέ πια αυτό το θέμα στην επόμενη θητεία. Να δούμε τι θα κάνει το πρόγραμμα δράσης. Αυτό να συζητάμε. Ευχαριστώ κύριε Κάσμαν για τη δέσμευσή σας αυτή και το στένωση. Κυρία Κώστα παρακαλώ. Νομίζω ότι είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι η πρακτική αυτή του ακροτηριασμού των γυναικείων και γενετικών οργάνων πρέπει να καταπλημεθεί σε δύο επίπεδα. Το πρώτο, το υπενθύμησε ο κ. Κάσμαν και άλλοι συνάδελφοι τη ομάδα μου των σοσιαλιστών και δημοκρατών, αλλά κάτι που μας βρίσκει σύμφωνος όλου μέσα από το ψήφισμα, είναι να υπάρξει νομοθεσία και συντονισμό ε, σύγκληση των, Ευρωπα... των εθνικών νομοθεσιών, καθώ και ευρωπαϊκή νομοθεσία σε κάποιες χώρες μόνο οι ανήλικοι προβλέπεται να προστατεύονται, ενώ σε άλλες δεν υπάρχει ούτε καν... Μάλλον σε άλλες είναι πολύ πιο σοβαρές οι ποινές και η απαγόρευση, όπως στην Ιταλία. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει συνεργασία, όπως σωστά είπε προηγουμένως πριν από λίγο ο Επίτροπος. Η Ευρώπη θα πρέπει να στείλει ηχηρά μηνύματα με... όταν προβλέπει συμφωνίες με διμερείς με διάφορες χώρες, διότι η εκστρατεία, η ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο σύνθημα που έχουμε ε, προβλέψει, στο more for more, περισσότερα για περισσότερα στις συνεργασίες με χώρες, όχι μόνο της Αφρικής. Ε, αλλά όπως είπε προηγουμένως και η κυρία Ματέρα, ε, σε χώρες όπως η δική μας, με σοβαρές εκστρατείες, με ένα δωρεάν νούμερο, υπάρχουν ακόμη κορίτσια σε οικογένειες που αποβάλλονται σε αυτού του είδους την βαρβαρότητα. Γι' αυτό λοιπόν στην Ευρώπη να μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς υπάρχουν ακόμη κοινότητες που θεωρούν αυτό το, ε, αυτή την πρακτική ως ένα τελετουργικό περάσματος ε, στην, από την εφηβεία στην ελληνική ζωή. Θα πρέπει λοιπόν στα σχολεία να υπάρξει εκπαίδευση, κάτι που ακόμα δεν έχει καλυφθεί επαρκώς. Ευχαριστούμε ο κύριος Κοφεράτη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ο ακροτηριασμό των γυναικείων γενετικών οργάνων, όπω σωστά υπόθηκε, είναι μια από τι χειρότερε μορφέ βία κατά των γυναικών είναι πραγματικά αποτρόπε και ιδίω κατά των ανήλικων γυναικών. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστεί με όλα τα μέτρα που, που έχουμε στη διάθεσή μα. Ε, είναι σημαντικέ οι δράσει που έχουν αναλυθεί ω τώρα, αλλά δεν είναι επαρκή. Νομίζω ότι χρήσιμο θα ήταν, όπω είπε προηγουμένω η συνάδελφο Κώστα, να δράσουμε και στο επίπεδο το πολιτιστικό. Δεν είναι δικαιολογία ότι πρόκειται για παράδοση, πρόκειται για μια βάρβαρη, απαράδεκτη πρακτική κατά των γυναικών. Πρέπει να ξεκινάμε λοιπόν από τα σχολεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε φορά που ε, εκπονεί μια πολιτική που αφορά τη γειτονία ή την ε, ε, οποιοδήποτε άλλο σκέλος της πολιτικής σα θα πρέπει να προβλέπει και ποινές για την ε, εξάσκηση της πρακτικής αυτής και εφόσον θέλει να διδοθούν τα βασικά ανθρωπίνα δικαιώματα, τα θεμελιώδη ανθρωπίνα δικαιώματα. Πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ανηλίκων και γυναικών. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να το αντιμετωπίσουμε αυτό και σε πολιτιστικό επίπεδο. Πρόεδρο, ευχαριστούμε κύριε Κοφεράτη. Και τώρα κυρία Τόμσεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε κύριε Επίτροπε. με την πρόφαση ότι είναι θρησκευτική και πολιτιστική παράδοση συνεχίζεται ο κροτηριασμός και στην Ευρώπη ακόμα. Περίπου 500.000 στην Ευρώπη ε, έχουν υποστεί και ε, σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες. 180.000 ε, γυναίκες και κορίτσια κινδυνεύουν στην Ευρώπη να υποστούν αυτό τον ακροτηριασμό. Είναι ε, μια από τις ε, πιο κατάφορες παραβιάσεις ε, ανθρωπίνων και γενικών δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει κανένας ιατρικός λόγος για να απομακρύνονται αυτά τα γεννητικά όργανα και συνήθως γίνεται αυτό χωρίς αναισθητικό με φρικτές συνθήκες υγιεινής. Είναι βαρβαρότητα, απανθρωπιά και αντιτίθεται και στις ε, θεμελιώδεις αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ένωση. Γι' αυτό καλωσορίζω την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ε, καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο του ακροτηριασμού και είναι καλή η μηδενική ανοχή που διακηρύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλό είναι όμως ε, να εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη, τα οποία οφείλουν να τα εφαρμόσουν. Χρειάζεται νομοθεσία, χρειάζεται πρόληψη ε, της βίας κατά των γυναικών, μια νομοθεσία που να ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να απαγορεύεται για να μπορέσουμε να εξαλείψουμε αυτό το φρικτό φαινόμενο. Ευχαριστώ κύριος Μέλτσερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με τη μαζική μετανάστευση από χώρες ε, εκτός της Ευρώπης έχουμε και τέτοια προβλήματα. Φόνους τιμής ή ακροτηριασμούς γενικών, γενικών οργάνων. Ε, πάνω από 20 χρόνια αυτό θεωρείται ε, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι εισεγόμενα φαινόμενα αυτά. μέχρι τώρα δεν έχουμε πρόοδους. Η ευαισθητοποίηση των υγειονομικών, η βοήθεια, οι συμβουλές, η συνεργασία ιατρικής αστυνομίας και δικαιοσύνης θα βοηθούσε πάρα πολύ. Πολλές μετανάστριες όμως ε, υφίστανται αυτό τον ακροτηριασμό όταν επιστρέφουν στις χώρες τους και δεν μπορούν οι υπεύθυνοι να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης όταν η πράξη αυτή έλαβε χώρα σε μια χώρα που δεν διώκεται ποινικά. Είναι έσχος που είναι 500.000 τα θύματα στην Ευρώπη και μέχρι σήμερα ε, δεν ε, έχουν ε, υπάρξει παρά μόνο πολύ λίγες διώξεις, μια χούφτα. Θα πρέπει επιγόντως να αλλάξει αυτό. Ευχαριστώ. Είμαστε στη δικασία Catch the τώρα. Η κυρία Πρέντεργαστ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, κάθε 11 δευτερόλεπτα ένα κορίτσι κάπου στον κόσμο αυτοτηριάζεται. Είναι μια βάρβαρη πρακτική. Η εκτομή των γενετικών οργάνων, η εκτομή της η ολοκληρωτική ε, εκτομή των γεννητικών οργάνων, με κομμάτια γυαλί ή ψαλίδια, ε, με ελλειπείς συνθήκες υγιεινής, είναι επικίνδυνη. Πολλές φορές το δέρμα που μένει αφού ε, γυναικτομή του γενετικού οργάνου, αιμορραγή και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος υγείας ή θανάτου. Ε, μιλάμε για μια μορφή βασανιστηρίου πάνω από 125 εκατομμύρια ε, γυναίκες. Είναι τραγικό να προσπαθεί μια τέτοια γυναίκα να ε, γεννήσει ένα παιδί. Ε, είναι φρικτή η αντίδραση των γυναικών αυτών όταν ε, γεννήσουν κορίτσι και για πραγματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πραγματικά μια πολύ καλή ευκαιρία σήμερα να φωτίσουμε λίγο τις φρικιαστικές πτυχές αυτού του φαινομένου. Ευχαριστούμε κύριε Μπένιον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μια γραπτή ερώτηση είχε απευθυνθεί προς τον Επίτροπο, παρόμοια με το προφορική ερώτηση σήμερα, όταν ένας ψηφοφόρος από το Μπέρμιχαμ ε, αναρωτήθηκε τι συμβαίνει με το φαινόμενο αυτό. Η κυβέρνηση συνασπισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο βέβαια έχει θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση αυτής της αποτροπής πρακτικής μια πρακτική που είναι απαράδεκτη. Απαράδεκτη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και επηρεάζει χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια σε όλη την Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω, γιατί δεν έχει κάνει περισσότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τους εταίρους της. Και τι δράσεις αναλαμβάνονται στα κράτη-μέλη για να καταπολεμηθεί αυτός ο κριτηριασμός, λόγω χάρη για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ή για το να φτάσουν ε, οι αυτές στις όπου τόσο πολύ απαντάται πρακτική αυτή. Ευχαριστώ κύριε Μπένιον. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση και το Κατδιάι. Ο λόγος στον κύριο Φίλε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να σα ευχαριστήσω που προβλέψατε τη συζήτηση για τον ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην ημερήσια διαταξή σήμερα. Κανένα κορίτσι δεν θα πρέπει να έχει αυτή την τραυματική εμπειρία, μια κατάφορη παραβίαση των θεμελιωδών τη δικαιωμάτων. Ευχαριστώ το Ευρωκοινοβούλιο και την ε, Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων για την αφοσίωσή του στην καταπολέμηση τη παραβίαση των, των δικαιωμάτων των γυναικών και του φαινομένου αυτού, τον εκατηρισμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Κάθε μέρα μια γυναίκα βιάζεται, ε, πέφτει θέμα ξυλοδαρμού, ή βασανίζεται στην Ευρώπη γιατί απλώ είναι γυναίκα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ε, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε το γεγονό ότι εκατομμύρια νεαρέ γυναίκε υποβάλλονται στον εκτελεσμό των γενετικών του οργάνων ε, ετησίω. Ε, κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή του και εάν επιζήσουν ζουν τραυματισμένες με κίνδυνο αναπηριών ή πολύ επικίνδυνων τοκετών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ε, δρά για την ενημέρωση των γυναικών και όλων και την ανάληψη των δικαιωμάτων των γυναικών, την προστασία τους καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλειών για την αποτροπή αυτού του ε, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει στοχοθετημένα και με στόχο τα αποτελέσματα προγράμματα ώστε τα κράτη-μέλη να πετύχουν περισσότερη πρόοδο στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Θα πρέπει οι γυναίκες να μπορούν να προσφύγουν στην ευρωπαϊκή ε, νομοθεσία και τις αρμοδιότητες της Ένωσης για να προστατευθούν. Ε, είναι πολλά τα κατημέλη που πρέπει να ανελάβουν εδώ δράση. Τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών αποτελούν μέρος των συζητήσεων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης όταν προβλέπεται ο προπολογισμό και τα κονδύλια που θα, ε, θα απευθυνθούν στην συνεργασία με μια τρίτη χώρα. Όμως εδώ δεν μιλάμε μόνο για μια μονομερή δράση αλλά για μια παγκόσμια συμφωνία. Οι εμπορικές μας συμφωνίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν να κάνουν και με τα συμφωνίες πλαίσιο που λειτουργούν ως πρότυπο για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Και όλα αυτά εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των συμφωνιών ε, συνεργασίας. Εκεί πάντοτε υπάρχει μια ρήτρα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο που καθορίζει τις σχέσεις μας με την τρίτη χώρα και ε, αποτελεί και έναν βασικό πυλώνα συνεργασίας, ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, ας συνεχίσουμε την στενή μας συνεργασία για το θέμα αυτό και ας εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία που μας παρουσιάζεται ώστε να μπορέσουμε να προβάλλουμε τα δικά μας επιχειρήματα. Θα συζητήσω και με τη συνάδελφο Ρέντινγκ σε ό,τι αφορά τις χρήσιμες προτάσεις σας ε, ιδίως αυτή της κυρίας Χολ προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φίλε. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει στη συνέχεια. Στι 12 το μεσημέρι βάσει των προτάσεων ψηφίσματο. Ακολουθεί τώρα προφορική ερώτηση Ναϊάδε 2, ένα πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοεία. Αποουσιάζει ο κύριο